Εδώ τελειώνουν λοιπόν οι ψηφοφορίες και περνάμε τώρα στις δηλώσεις, επεξηγήσεις μάλλον ψήφου. Θα περιμένω κάποια στιγμές για να βγουν οι συνάδελφοι από την αίθουσα. Ενώ οι συνάδελφοι που δεν ενδιαφέρονται εξέρχονται τις αιθούσεις, ξεκινάμε με τις επεξηγήσεις ψήφου. για την πρόταση ψηφίσματος ε, για την ένσταση με βάση το άρθρο 106, δηλαδή την ανανέωση της έγκρισης της ε, δραστήριας ουσίας γλυφωσάτης, Ζήτησε να μιλήσει η κυρία Ρόζα Νταμάτο. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρο. Εδώ κάναμε δημοκρατική έκκληση στη σεβασμό της αρχής της προφύλαξης που δεν εφαρμόζεται από την Κομισιόν και μάλιστα αντί να επικρατήσει η υποστήριξη του δημοσίου συμφέροντος ε, θυμίζουμε ότι η Μονσάντο έχει δηλώσει ότι αυτά είναι θεμελιώδη για την αρνητική γνωμοδότηση όσον αφορά το κατά πόσο είναι καρκινογόνα ή όχι η ουσία γλυφοσάτη τι, διαβα... τι είδαμε και τι πετύχαμε, κάτι που δεν ξέρουμε καν πώς θα λειτουργήσει. Αυτό που επαιτούμε είναι οι μελέτες να είναι δημόσιες, δεν το λέω εγώ, αλλά το άρθρο του κανονισμού για την εμπορευματοποίηση των φυτογενομικών προϊόντων. Ο Επίτροπος ατριοκαρίτης έχει ευθύνε. Ε, αυτή η διαδικασία δεν μπορεί και δεν πρέπει να προχωρήσει. Γι' αυτό και ζητήσαμε ένα ψήφισμα τελείως τρελό, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε την ανανέωση της ε, αδειοδότησης της γλυφωσάτης για ακόμα 7 χρόνια. Είναι πραγματικά ασυνείδητο από πλευράς ε, όλων εδώ να έχουν υπερψηφίσει τον μη σεβασμό της υγείας όλων μας των πολιτών. Ε... Αν οι συνάδελφοι που βγαίνουν, βγαίνουν λίγο πιο ησύχω, ε, θα ήταν καλύτερο και θα ήταν και έδειχναν σεβασμό στους ομιλητές. Ναι, Μάκερ είναι εδώ. Δεν είναι. Λόμπε Λόπες Βερβέγιο. Τσε. Είναι, δεν είναι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, όσον αφορά την ε, συζήτηση για τον γλυφοσάρτα, τους εχθρούς και τους ε, φίλους της πρόοδου υπάρχει ένα κέντρο διεθνών ερευνών για τον καρκίνο το οποίο ταξινόμησε το γλυφοσάτ ως ε, καρκινογόνο στη βάση της αρχής της πρόληψης και το κείμενο της ε, έγκρισης η Κομισιόν δεν μπορεί να προχωρήσει σε μια άμεση έγκριση. δεν ε, μπορεί να γνωρίσει βεβαίως τις κινδύνους για, υγείας, για την υγεία. Ε, πολλές χώρες έχουν αντιταχθεί ε, σε μια έγκριση. Εμείς από την Ενωτική Αριστερά έχουμε αντικαταστήσει σε πολλούς δήμους το γλυφοσάτ με μεθόδους λιγότερες επικίνδυνες και επιμένουμε ότι υπάρχουν κάποιες εναλλακτικές λύσεις. Δεν ε, ισχύει το επιχείρημα το οποίο ευνοεί την χρήση αυτών των ε, χημικών φαρμάκων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Στην ε, Ανατολική Αγγλία λαμβάνω εκατοντάδες ε, mail από τους καλλιεργητές για το γλυφοσάτ. Είναι το μόνο μέσο, λένε, που διαθέτουν για να ελέγξουν τις ε, ασθένειες και είναι πολύ σημαντικό για, την, για όπως είναι το κρυθάρι, το και κλπ. Ο αντίκτυπος για την απαγόρευση του γλυφοσάτ θα ήταν τεράστιος. Ε, πρέπει οι καλλιεργητές να παράγουν ε, τα προϊόντα για την διατροφή και μας λένε ότι το γλυφοσάτ δεν είναι πολυτέλεια, είναι απολύτως, ε, απαραίτητο. Ωστόσο, πολλοί ανησυχούν για τους κινδύνους υγείας και θα πρέπει να συνεχίσει η έρευνα. Οι σοσιαλιστές ζητούν παρόλα αυτά μια άμεση απαγόρευση τώρα. Εγώ διαφωνώ. Θα πρέπει να αφήσουμε τους καλλιεργητές και τους επιστήμονες να κάνουν ε, τη δουλειά τους και να δώσουμε ένα περιθώριο χρόνου έως ότου καταλήξουμε σε μια τεκμηριωμένη τοποθέτηση. Voilà. κυρία Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρο. Εγώ η ίδια είχα προτείνει από την ομάδα ENF να υπάρξει μια αντίρρηση στην ανανέωση τη έγκριση του γλυφοσάτη. Ήταν μια πρωτοβουλία που δεν έγινε δεκτή από τι άλλε πολιτικέ ομάδε που προτίμησαν να παρουσιάσουν ένα δικό του κείμενο. Παρ' όλα αυτά, είδαμε σήμερα ότι υπάρχουν μεγάλε διαφορέ και στο εσωτερικό των μεγάλων πολιτικών κομμάτων. Εγώ λοιπόν ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κατανοήσει ότι προτείνοντας την συνέχιση της έγκρισης του γλυφοσάτ έχει υπερβεί τις εξουσίες της. Οι επιστημονικές μελέτες και τα στοιχεία του Διεθνούς Κέντρου Έρευνας για το Καρκίνο πρέπει να μας κάνουν να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί σε σχέση με ένα προϊόν το οποίο είναι πανταχού παρόν και ενδεχομένω καρκινογόνο. Αυτό θα πρέπει να είναι το κέντρο της ε, άποψης της Κομισιόν όπως τόνισε και η διαμεσολαβήτρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούμε να παραπέψουμε σε μια ημερομηνία άγνωστη την δημοσίευση για στοιχεία που είναι τα, τα συνά, ε, συνέκδοχα του γλυφοσάτ και μπορούν να αυξήσουν την τοξικότητα του προϊόντος. Πρέπει λοιπόν να παρουσιαστούν όλα τα στοιχεία αυτά που ζητάει η αντίληψή μας. Η κυρία Τόρες Μαρτίνες, για ένα λεπτό. Παρακαλώ καταψηφίσαμε δεδομένου ότι οι τροπολογίες που εγκρίθηκαν δεν ανταποκρίνονται στο αποτέλεσμα των συζητήσεων που είχαμε στην αρμόδια επιτροπή. Είναι θέμα ανευθυνότητα να ζητήσει η ανανέωση του γλυφοσάτη να λάβει χώρα για 7 χρόνια. Υποδέμω ζητά από τις αρμόδιες αρχές να εφαρμόσουν την αρχή της πρόληψης η έκθεση της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγεία τόνισε ότι κατά πάσα πιθανότητα είναι καρκινογόνο για τους ανθρώπους το γλυφοσάτ. Έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία τροφιμικής ασφάλειας έχει άλλα συμφέροντα που υποκρύπτονται αυτής γιατί έφτασε σε αντίθετα συμπεράσματα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε λοιπόν να υπάρχει εμπορευματοποίηση στην Ευρώπη μιας ουσίας που έχει τέτοιους κινδύνους που χρησιμοποιείται σαν λίπασμα για τα χωράφια μας και καταλήγει στα τρόφιμά μας και θέτει σε κίνδυνο το έργο των γεωργών και των κτηνοτροφών. κτηνοτροφών. Δεν μπορούμε να παίζουμε με την υγεία των λαών μας. Ο κύριος Γιάρ. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, φαντάζομαι ότι αν συμφωνούμε στην πολιτική για μια διαδικασία θα πρέπει να σεβαστούμε αυτή τη διαδικασία μέχρι τέλους και να αποδεχθούμε επίσης και τα αποτελέσματα. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια επιστημονική ειδική αξιολόγηση ε, ε, και η Ευρωπαϊκή ΕΦΣΑ έλαβε υπόψη στα αποτελέσματα της έρευνας και κατέληξε σε κάποιες αποφάσεις και θεωρώ ότι η σημερινή απόφαση σήμερα πραγματικά δικαιολογεί αυτή την ε, ε, τεκμηρίωση. Θα επιθυμούμε να ορίσουμε επακριβέστερα την εφαρμογή της χρήσης του γλυφοσάτ και θέλουμε να συνεχίσουν οι επιστημονικές έρευνες ιδιαίτερα όσον αφορά την μακροπρόθεσμη δράση του γλυφοσάτ. Ε, θεωρώ ότι ήταν μια σωστή απόφαση στη βάση μιας επιστημονικής ε, τεκμηρίωσης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ ε, επέλεξα να δω το ε, ποτήρι κατά ίμιση γεμάτο. Ε, σε σχέση με την ανέωση της έγκρισης του γλυφοσάτ ε, για 15 έτη, όπως το επιθυμούσε η Κομισιόν, ε, το Κοινοβούλιο έδειξε ότι στέκεται στο πλευρό των πολιτών. Γιατί είναι ο δικός μας, εναπόκειται σε εμάς πολιτικούς να πάρουμε τις αποφάσεις. Βεβαίως οι ειδικοί καλούνται να προβούν σε επιστημονική τεκμηρίωση. Εδώ πέρα οι γνώμες διχάζονται, αλλά το δικό μας ε, ε, μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Λέμε ναι για την ε, ανανέωση της έγκρισης του γλυφοσάτ για 15 χρόνια. Τα, η διάρκεια των 7 ετών που ψηφίστηκε παραμένει αρκετά μεγάλη και θα πρέπει στη συνέχεια να ψηφιστεί και να προταθεί ένα νέο κείμενο το οποίο θα υποβληθεί στις χώρες μέλη. Ο κύριος Πόσελ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ ψήφισα κατά της πρότασης Κομισιόν για την ανανέωση της έγκρισης για τα επόμενα 15 χρόνια. Γιατί είμαι πεπισμένος ότι από τη στιγμή που υπάρχουν σαφείς επιστημονικές ενδείξεις που διαμφισβητούν την ε, ασφάλεια αυτής της χημικής ουσίας δεν μπορούμε να είμαστε ανεύθυνοι και να παρατείνουμε την έγκριση του προϊόντος αυτού. Ήταν σαφή τα στοιχεία που μας έδωσε η Επιτροπή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την κακοινογενή μορφή αυτού του προϊόντος. Τόνισε η Επιτροπή αυτή ότι μπορεί να είναι καρκινογόνο και ενδεχομένω έχει ήδη καρκινογόνο αποτέλεσμα στους ανθρώπους. Αυτή τη στιγμή παίζουμε παιχνίδια με την υγεία των πολιτών μας. Είναι πολύ θετικό λοιπόν το ότι η Κομισιόν δεν πήρε τα 15 χρόνια που, πήρε, που ήθελε να πάρει για την παράταση. Όσο παραμένουν φόβοι για τον ε, καρκινογενή ε, χαρακτήρα αυτής της ουσίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα έπρεπε να επιτρέπει τη χρήση του. Θα έπρεπε να έχει ε, την πρωτοκαθεδρία η δημόσια υγεία. Ε, τόσο δύσκολη ε, διαδικασία δείχνει, εδώ στο Κοινοβούλιο δείχνει ότι δεν λειτουργήσε η, σωστά η διαδικασία και ότι κάτι πάει στραβά. Ε, υπάρχουν ε, βάσιμοι φόβοι ότι είναι καρκινογόνα αυτή η ουσία και μάλιστα μείγματα γλυσοφωσάτης με άλλες ουσίες μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρούς κινδύνους για την υγεία, για τους πολίτες αλλά και για τους αγρότες. Η Γαλλία μάλιστα αποφάσισε να απαγορεύσει τα ε, σκευάσματα με γλυφοσάτη. Δεν, παρόλα αυτά η Κομισιόν θέλει να παρατείνει την άδεια. Πρόκειται για μια παράλογη θέση όταν διακυβεύεται η υγεία των πολιτών. Η Κομισιόν αντίθετα θα έπρεπε να παρουσιάσει μια ε, μελέτη ανεξάρτητη με βάση όλα τα διαθέσιμα στοιχεία σε σχέση με την ε, ε, το κατά πόσο είναι καρκινογόνα και τους επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Ευχαριστώ. Και κυρία Εύη, ευχαριστώ. Το Ευρωκοινοβούλιο είχε τη δυνατότητα να εκφράσει μια έντονη πολιτική θέση κατά της ανανέωσης της άδεια του γλυφοσάτης που είναι ζανεκτόνο και που θεωρείται βλαβερό και καρκινογόνο. Ε, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξέρουμε ότι έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει και να υιοθετήσει πράξεις και διατάξεις αυτόνομα. Όμως εδώ είναι σημαντικό να εκφραστούμε και είναι πραγματικά κρίμα ε, αυτό που συνέβη. Το κίνημα των πέντε αστέρων ήταν ανάμεσα στους μεγαλύτερους υποστηριχτές ε, της ε, υιοθέτησης αυτής της πρότασης και τελικά χρειάστηκε να το καταψηφίσουμε. Μάλιστα μετατρέψαμε μια πρόταση ενστάσεως σε, μια πρόταση παράτασης για άλλα 7 χρόνια. Η υγεία των πολιτών όμως δεν μπορεί να ακολουθεί μόνο τις εμπορικές ευκαιρίες των μεγάλων πολυεθνικών. Ευχαριστώ. Ο κ. Σον Κέλλη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι ήταν λογική αυτή η συμβαστική λύση να εγκρίνουμε για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα. Δεν μπορούμε να βασιζόμαστε σε στοιχεία τα οποία δεν είναι ασφαλή. Το να πούμε κάτι ότι είναι πιθανός καρκινογόνο είναι σοβαρό. Γι' αυτό περιορίσαμε σε 7 χρόνια. Υπάρχουν και άλλες πτυχές ε, που αφορούν το θέμα αυτό. Λοιπόν, πρέπει να έχουμε τα απαραίτητα στοιχεία για να εξασφαλίσουμε ότι αυτό το προϊόν είναι απόλυτα ασφαλές για τους ανθρώπους γιατί αυτό το προϊόν περνάει και στην τροφιμική αλυσίδα. Νομίζω ότι η απόφαση αυτή είναι θετική γιατί επιτρέπει στους γεωργούς να συνεχίσουν να το χρησιμοποιούν χωρίς να υπάρξει σημαντική διαταραχή στην γεωργία και έτσι μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα να ξέρουμε τι ακριβώς σημαίνει, σημαίνει και να διαβιβλώσουμε τους πολίτες μας ότι όλα αυτά που έχουν στα τρόφιμά τους είναι απόλυτα ασφαλή. Ένα λεπτό κύριο Μάμικινς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ένα από τα κύρια προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε είναι ότι το glyphosate δεν είναι επιλεκτικό σκοτώνει τα παράσιτα, τα ζυζάνια, αλλά και τους μύκητες και τα φύκη και άλλα ζωντανά όντα και είναι κάτι το αρνητικό για τη βιοποικιλότητα. Κατανοώ ότι το σχέδιο της Κομισιόν δεν προβλέπει να δεν έχει σαν αποτέλεσμα την, την ε, εξασφάλιση της ανθρώπινης υγείας. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει το ταχύτερο δυνατό μια μελέτη των ε, επιπτώσεων του γλυφοσάτ για, ε, για τον καρκινογόνο ρόλο του και τον αντίκτυπό του στο ενδοκρινικό σύστημα των ανθρώπων. Πιστεύω λοιπόν ότι η Κομισιόν θα πρέπει να δημοσιεύσει πλήρως τα στοιχεία τα οποία πετέλεσαν τη βάση της αίτησης της για ανανέωση. Ο Μάρκ Θαραμπέλα, κύριε Πρόεδρε, ψηφίσαμε για μία αντίρρηση του Κοινοβουλίου σε σχέση με την ανανέωση που ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτή την επικίνδυνη ουσία των γλυφοσάτ. Η Κομισιόν ήθελε για 15 χρόνια ζήτησε κάτι τέτοιο. Ήταν ανεύθυνο αυτό το οποίο κάναμε να ψηφίσουμε για μία αντίρρηση και μετά να πούμε ότι θέλουμε 7 χρόνια να συνεχιστεί η έγκριση. Δεν μπορούμε λοιπόν να ε, κάνουμε μία απόφαση αυτού του είδους όπως η τροπολογία 11 του ΕΛΚ η οποία θέλει να επιτρέψει την, ε, την ε, έγκριση για 7 χρόνια. Είναι σαν να παίρναμε ένα ποταμό και να σταματάμε στη μέση του ποταμού. Είναι κάτι το οποίο αλλοιώνει το μήνυμα το οποίο ε, θέλαμε να δώσουμε. Γι' αυτό εμείς ως Βέλγοι Σοσιαλιστές κρατήσαμε στάση αποχής. Τονίσαμε ότι ήταν σημαντική αυτή η απόφαση, αλλά δυστυχώς χάθηκε η δύναμη του μηνύματος με το να ζητήσουμε την έγκριση για 7 χρόνια. Ο κύριος Πολ Τσακ. Ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ. Η γνώμη μου ε, για αυτό το θέμα ήταν υποεξέλιξη και άλλαξε από την τελευταία φορά και γι' αυτό και ελεύθερα επέκρινα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δεν μας έδωσε αρκετά επιστημονικά στοιχεία. Από την άλλη πλευρά η Γεωργή μου εξήγησε ότι από τη μια πλευρά η γλυφοσάτη μπορεί να είναι καρκινογόνα, από την άλλη πλευρά όμως το ίδιο ισχύει για τις εκπομπές των αυτοκινήτων και τα αυτοκίνητα δεν απαγορεύονται. Γι' αυτό και ε, συμφώνησα με τη συμβιβαστική πρόταση που κατετέθη στο σώμα και που κρίθηκε. Επίσης άλλαξα την γνώμη, άλλαξε η γνώμη μου από την ε, τελευταία ολομέλεια όπου είχα γιατί μπόρεσα να μελετήσω την άποψη των γεωργών μας. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι αυτή η περίοδος θα πρέπει να ε, χρησιμοποιηθεί για να μελετήσουμε όχι μόνο την γλυφοσάτη αλλά και όλες τις άλλες ουσίες, χημικές ουσίες. Αυτή ήταν τελευταίος ο για την γλυφοσάτη και περνάμε στην έκθεση Καλνιέτε όπου έχει ζητήσει το λόγο η κυρία Μορβάη για ένα λεπτό παρακαλώ. Αγαπητοί Ευρωπαίοι πολίτες, θα έπρεπε να έχουμε επέγνωση σχέση με το τι συμβαίνει στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο. Ε, υπάρχουν πράξεις επιθετικότητας κατά ορισμένων εθνών και της ε, διάθεσής τους. Αυτή η έκθεση συνιστά μια μαζική επίθεση υπό την έννοια αυτή και ενώ η παγκόσμια διακυβέρνηση θα πρέπει να ενισχυθεί και αναφέρεται αυτός ε, ρητός ε, στόχος θα μπορούσα να σας αναφέρω σχετικά πολλά παραδείγματα που δείχνουν ότι ο στόχος είναι να προωθηθούν διάφορα προϊόντα στην παγκόσμια αγορά και να προστατευτεί η σταθερότητα του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος. όλες οι συμβάσεις για τον ενεργειακό εφοδιασμό και την υπογραφή αυτών των συμβάσεων η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να έχει την ε, αρμοδιότητα. Ο κύριος Γιάρ, κύριος Γιάρ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κατ' ουσία η έκθεση αυτή περιλαμβάνει τέσσερα σημεία. Το πρώτο σημείο αφορά την ε, περάσπιση των ευρωπαϊκών χωρών δηλαδή είναι αναγκαίο να ενισχυθεί αυτή η δυνατότητα των χωρών. Δεύτερον, πρόκειται για την ε, σταθεροποίηση της άμεσης γειτονία της Ευρώπης και αυτό είναι σωστό. Τρίτον, το ζητούμενο είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να κατατείνει ε, περισσότερο στην κατεύθυνση του να θέτει τους κανόνες, δηλαδή να μην παρατηρεί αλλά να επηρεάζει ενεργά τις εξελίξεις. Και τέταρτον, και αυτό το σημείο θεώρησα εγώ ότι είναι ιδιαίτερο ενδιαφέρον, το ζητούμενο είναι να υπάρξει μια ρήτρα αναθεώρησης, δηλαδή κάθε πέντε χρόνια αποκινούμε τα Εθνικά Κοινοβούλια και τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συζητούμε εν σχέση με το πώς θέλουμε να συνεχίσουμε τις εργασίες μας σε αυτό το χώρο. Άρα λοιπόν η έκθεση αυτή είναι θετική και δεν μπορούμε παρά να την υπερψηφίσουμε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πόσπιση, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ υπερψήφισα τελικά παρά το γεγονός ότι κάποιες ιδέες οι οποίες αφορούσαν την αμυντική ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρούσα ότι είναι υπερβολικές γιατί λέει παραγωγός χάρη ότι το ΝΑΤΟ θα πρέπει να είναι αρμόδιο για την να είναι ο κύριος ε, σύμμαχός μας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ε, οι επίσης οι εκεί που λένε ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες και να υπερβούν το 2,5% του ΑΕΠ τους. Δεν μπορούμε λοιπόν να θεωρούμε ότι η άμυνα είναι κάτι που δεν έχει καμιά σχέση για με εμάς και μπορούμε να δαπάνουμε τα χρήματα αυτά σε άλλα θέματα εκτός άμυνας. Έχω αμφιβολίες όμως για την κοινή Ευρωπαϊκή Ένωση για τα αμυντικά θέματα. Καλύτερα να δουλεύουμε με τον ΝΑΤΟ και όχι να κάνουμε παράνο, παράλληλες στο Μεσοκύριο και Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ έχω ανάμεικτα αισθήματα χαράς και λύπης σε σχέση με αυτήν την πρόταση. Είναι γεγονός ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και δεκαετίες έχουμε παίξει ένα σημαντικό όρπλο σε παγκόσμιο επίπεδο. Μιλάμε και για το στρατιωτικό χώρο. Έχουμε τα καθήκοντά μας μέσα στο ΝΑΤΟ και τα κράτη-μέλη έχουν ένα δυναμικό το οποίο δεν χρησιμοποιείται επαρκώς, αλλά συγχρόνως είναι ανάμεικτα τα θέματα αυτά. Πρέπει να δαπανίσουμε το 2% του ΑΕΠ μας για στρατιωτικούς λόγους να ενισχύσουμε τη σχέση μας με τους Αμερικανούς γιατί παίρνουμε απειλέ από τα ανατολικά και επομένως λόγω αυτών των ανάμεικτων συναισθημάτων καταψήφισα την έκθεση γιατί δεν νομίζω ότι είχε προετοιμαστεί όρθα. Ευχαριστώ κύριος Πόλτσακ. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ υποστήριξα αυτή την έκθεση για πολλούς λόγους. Καταρχήν πιστεύω ότι το μοντέλο μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής ε, γειτονίας είναι θετικό και περιγράφεται και καλά. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες να είναι εταίροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ωστόσο το μοντέλο αυτό της ευρύτερη γειτονία, της ευρωπαϊκής θα πρέπει να ενισχυθεί. Έστω και αν μια χώρα δεν μπορεί ακόμα να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θεωρώ ότι περιγράφεται αυτό όλο πολύ καλά στην έκθεση αυτή. Επίσης είμαι υπέρ μιας ενίσχυσης και εμβάθυνσης της αμυντικής μας στρατηγικής περιλαμβάνοντας και την δικτύωση δική, τις δικές μας ε, αμυντικές ε, ομάδες ε, και ομάδες ασφαλείες παρόλο που έχουμε το Βερολίνο 1 και Βερολίνο 2 που δίνει τη δυνατότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση να χρησιμοποιεί μονάδες του ΝΑΤΟ. Παρ' όλα αυτά αυτό δεν είναι εφικτό για το μέλλον. Θα πρέπει να έχουμε τις δικές μας αμυντικές και στρατιωτικές μονάδες και δυνατότητες. Σήμερα εστιάζομαι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 στον ε, έλεγχο μιας ε, ευρείας αμυντικής ε, στρατηγικής. Ωστόσο, με καταπλήσει το γεγονός ότι αυτή η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγινε πολύ κοντά στην ημερομηνία του Brexit και ξέρουμε πως επίμαχνε το θέμα αυτό στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εγώ καταξήφισα κάθε θέμα το οποίο συνδέεται με την διεύρυνση της, ευρωπαϊκής, της αμυντικής και στρατηγικής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, δεν είναι ενδεδειγμένη η στιγμή για να γίνει κάτι τέτοιο και εγώ δεν μπορώ να υποστηρίξω ε, την ευρωπαϊκή ε, παρέμβαση και την αύξηση του στρατιωτικού ελέγχου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρία Μακοβέη, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το 2013 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έθεσε σαφούς, σαφείς στόχους για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτα απ' όλα σε σχέση με ένα καθεστώς προμηθειών και επίσης την ενίσχυση των βιομηχανικών ικανοτήτων που έχουν να κάνουν με τον αμυντικό χώρο και τρίτον για την παρακολούθηση των προμηθειών στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας. Αλλά η Κομισιόν δεν έχει εκπληρώσει αυτούς τους στόχους και αυτό σημαίνει απώλεια ανθρωπίνων ζώων ο Ευρωπαϊκός στρατός θα πρέπει να γίνει το ταχύτερο δυνατόν πραγματικότητα. Πρέπει να ενισχύσουμε και τις σχέσεις μας με τον ΝΑΤΟ, την εταιρική μας σχέση και να καλύψουμε το κενό ασφαλείας που έχουμε στην περιοχή μας. Εάν υπήρχε κάποτε ένας χρόνος και μια εποχή αλληλεγγύης, είναι εδώ και τώρα να αγωνιστούμε για να προστατεύσουμε τις ζωές και την ελευθερία και την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εδώ τελείωσαν οι επεξηγήσεις ψήφου για την έκθεση Καλνιέτερ και πάμε στην έκθεση Μέζεριξ. Η κυρία Γιαρόκα για ένα λεπτό έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να εξηγήσω γιατί ε, απήχα δεν μπορούσα να καταψηφίσω το ψήφισμα γιατί συμφωνώ με τη βασική ιδέα της έκθεσης. Πράγματι, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια συνεκτική προσέγγιση, μια προσέγγιση με συνέπεια έναντι της ευρύτερης περιοχής αυτής για να μην στείλουμε συγκεχημένα μηνύματα στην κοινή γνώμη. Γι' αυτό δεν μπορούσα να την καταψηφίσω, αλλά δεν μπορούσα ούτε και να την υπερψηφίσω, διότι θεωρώ ότι το κείμενο δεν παρουσιάζει καθόλου συνοχή και καθόλου συνέπεια σε σχέση με τη δική μας θετική παράδοση. Έχουμε διαφοροποιήσεις των εθνών, των ε, πολιτισμών ε, και δεν έχουμε επαρκή σεβασμό προς τους εταίρους μας. Με την ιδιότητά μου λοιπόν τη συμμετοχή στην Επιτροπή Συνεργασίας ε, Ευρώπης-Ασίας προτείνω να έχουμε διατύπωση περισσότερο προς την κατεύθυνση του αμοιβαίου σεβασμού. Ευχαριστώ. Πώς πισιπίλ για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, στήριξα την έκθεση αυτή διότι πιστεύω ε, σε αντίθεση με τους προλαλήσοντες ότι πράγματι υπάρχει λόγος να ομιλούμε για ανθρώπινα δικαιώματα στην Νοτιοανατολική Ασία. Είναι μια περιοχή με πολύ ελπιδοφόρο μέλλον και πρέπει να συνεργαζόμαστε με την περιφέρεια την ευρύτερη. Ωστόσο, να μην μας ενδιαφέρει μόνο η οικονομία και η επιχειρηματική συνεργασία. Να υπογραμμίσουμε το ότι και τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν σημασία. Άλλωστε, το ότι συνεχίζονται οι συζητήσεις αυτές εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι κάτι το πολύ καλό και στην Τσεχία το ίδιο συμβαίνει. Έχουμε ένθερμες και τεταμένες συζητήσεις για τις σχέσεις μας με την Κίνα. Άλλωστε, ο Πρόεδρος μόλις επισκέφθηκε τη Τσεχική Δημοκρατία. Και θέλουμε να ξέρουμε η ύλη έχει σημασία ή ε, το άϊλο, το νοητό. Ποιο από τα δύο προτεύει. Πρέπει να συνεργαστούμε με αυτές τις χώρες, αλλά να εφιστήσουμε την προσοχή και στα υφιστάμενα προβλήματα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Κεντρική Ασία βρίσκεται αρκετά κοντά στην Ευρώπη σε σύγκριση με την Νότιο Αμερική, αλλά τη τελευταία δεκαετία δεν έχει λάβει την απαραίτητη προσοχή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λαμβάνοντας ε, υπόψη την ε, Προεδρία της Λετωνίας και την άποψη της Λετωνίας έχει αλλάξει η πολιτική ελαφρώς. Αυτή η περιοχή πολιτικά και οικονομικά έχει ε, ουσιαστικά επηρεαστεί από τη Μόσχα, το Πεκίνο, αλλά θα μπορούσαμε κι εμείς να κάνουμε τη δική μας συνεισφορά. Βλέπουμε ότι όλες οι χώρες έχουν τις δικές τους αρχές διακυβέρνησης και είναι πάρα πολύ παλιές και μάλιστα μπορούν να αναχθούν και στην εποχή που ανήκαν στη Σοβιετική Ένωση. Τώρα έχουμε την ε, πρόταση για την επιδημία του ιού πρόταση ψηφίσματος, παρακαλώ για ένα λεπτό. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως είπα κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την επιδημία του Ιουζίκα στην προηγούμενη Ολομέλεια, τώρα ε, ε, ουσιαστικά είναι εντελώς ε, απαράδεκτο αυτή η θεραπεία που δίνεται. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταχράται την κατάσταση των πληθυσών γυναικών μετά από δεκάδες χρόνια οι χώρες έχουν αντισταθεί στην πίεση των δυτικών οργανισμών για να επιβάλλουν αυτή την κουλτούρα του θανάτου και βλέπουμε τώρα πως οι γυναίκες στον αναπτυσσόμενο κόσμο αντί να λάβουν βοήθεια οδηγούνται στις αμβλώσεις. Οι έγκυες αντιμετωπίζουν ανασφάλεια και δύσκολες συνθήκες. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε αυτούς. Σας ευχαριστώ. Κυρία Μορβάη, για ένα λεπτό. <clears throat> Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Φυσικά υπερψήφισα την έκθεση αυτή. Πώς να ψηφίσει κανείς κάτι διαφορετικό άλλωστε. Ποιος δεν θα υποστήριζε μια τέτοια έκθεση. Ε, πρέπει όμως να βγάλουμε ορισμένα διδάγματα. Και έχω και κάποιες επιφυλάξεις. Το υπερψήφισα με βαριά καρδιά γιατί όταν μελέτησα το κείμενο έχω πρόβλημα. Ε, έψαχνα να βρω που κρύβονται τα συμφέροντα των πολυεθνικών φαρμακευτικών εταιριών ή ε, που είναι τα συμφέροντα των κυρίαρχων ε, μέσων ενημέρωσης. Παρουσιάζουν σωστά την κατάσταση ή όπως θέλουν εκείνα. Και τι γίνεται με αυτή την κουλτούρα ε, των ε, αμβλώσεων που θέλει ο δυτικός κόσμος να επιβάλλει και στον αναπτυσσόμενο. Όλα αυτά λοιπόν είναι κάποιες επιφυλάξεις που πιστεύω ότι είναι δικαιολογημένες και κάποιες απορίες που έχω και αμφιβολίες. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η πρόληψη και εκεί θα πρέπει να ποντάρουμε και όχι στις αυλώσεις. Από την άλλη έχουμε τα παγκόσμια συμφέροντα ε, των μεγάλων ομίλων, των μεγάλων εταιριών και οι άνθρωποι είναι εκτεθειμένοι και είναι έρμεα στα χέρια όλων αυτών των συμφερόντων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πόσπισιλ παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Αποφάσισα να πάρω το λόγο γιατί η ψηφοφορία δεν ήταν ονομαστική για το θέμα αυτό. Ήθελα λοιπόν να καταγραφώ στα πρακτικά εγώ θεωρώ αυτή την έκθεση πάρα πολύ σημαντική και γι' αυτό την ψήφισα. Εκ πρώτη όψεω μπορεί να φαίνεται ότι αυτό το πρόβλημα δεν αφορά την Ευρώπη. Παρ' όλα αυτά, αυτή είναι μια κοντόφθαλμη προσέγγιση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως παγκόσμιος δεν θα πρέπει να απορρίψει την διεθνή της ευθύνη. Γι' αυτό λοιπόν καλό είναι που υποστηρίζουμε με 10 επιπλέον εκατομμύρια ευρώ τη μελλοντική έρευνα. Δεν ξέρω αν θα φτάσουν αυτά τα χρήματα. Αν δεν επαρκούν, τότε θα πρέπει να αυξήσουμε αυτά τα κονδύλια και να προσπαθήσουμε να βρούμε περισσότερες πληροφορίες για τη σχέση μεταξύ του ιού και της δυσπλασίας του κεφάλου. Ευχαριστώ, κύριος Μαμίκης. Ευχαριστώ. Φυσικά, η εξέλιξη δεν ισχύει μόνο για τους ανθρώπους και οι μεταλλάσσονται συνεχώς και γίνονται όλο ένα και πιο επικίνδυνοι. Ο ιός Ζήκα είναι ένα από τα τελευταία παραδείγματα. Μία από τις μεγαλύτερες διαφορές είναι ότι έχει τεράστια επίπτωση στα έμβρια επίσης ε, πλήττει και τους ενήλικες. Άνθρωποι, πάρα, χιλιάδες άνθρωποι έχουν πληγεί ε, στην Νότια Αφρική και στην Νότια Αμερική, συγγνώμη στην Αφρική και στην Νότια Αφρική. Διαδίδεται ιός, λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψη, στήριξα την άποψη της Κομισιόν σε σχέση με τα 10 εκατομμύρια ευρώ για την έρευνα. και ζήτησα από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να ασχοληθούν με το θέμα. Σας ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στην κατάσταση στην Πολωνία. Μάρουση για δύο λεπτά. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, głosowaliśmy tutaj przed chwilą rezolucję w sprawie oceny. Κοιτάξτε, πριν από λίγο το ψήφισμα για την αξιολόγηση της κατάστασης στην Πολωνία σε σχέση με το κράτος δικαίου. Το περίεργο είναι ότι το ψήφισμα αυτό δεν λέει και πολλά στην ουσία του δεν συμβάλλει στην όλη συζήτηση για το κράτος δικαίου στη Πολωνία. Όμως λέει πολλά για την κατάσταση του κράτους δικαίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα. Η συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν δίνει στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δικαίωμα να ελέγχουν και να αποφασίζουν ε, για τις διάφορες πτυχές του κράτους δικαίου. Αυτό είναι εθνική εσωτερική αρμοδιότητα των κρατών μελών. Επομένως, Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει ότι δεν ενδιαφέρει καθόλου το κράτος δικαίου γιατί δεν τηρεί, δεν τηρεί και δεν σέβεται την νομοθεσία που έχει η ίδια εγκρίνει και ψηφίσει για τον εαυτό της. Νομίζω ότι έρχονται σε δύσκολη θέση τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Είμαι Πολωνός πατριώτης και ανέκαθεν προσπαθώ να με τα δικαιώματα της Πεολονία. Δεν μιλώ όμως τώρα ως Πολωνός πατριώτης, αλλά ως εκπρόσωπος της ε, πολιτικής ε, δεξιάς. και ως κάποιος που γνωρίζει πολύ καλά το κράτος δικαίου. Δεν θα ήθελε η Ευρωπαϊκή Ένωση να έρχεται σε αυτή τη δύσκολη θέση. Δεν θα πρέπει μόνο οι υπόλοιποι να συμμορφούνται με τους κανόνες, αλλά και εμείς οι ίδιοι στην Ευρώπη να γνωρίζουμε και να σεβόμαστε τη δική μας νομοθεσία. Αν θεωρούμε ότι είναι λάθος η νομοθεσία, ας την αλλάξουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά ας την τηρήσουμε προς το παρόν την ευρωπαϊκή νομοθεσία, ε, προτού απαιτήσουμε από τους άλλους να τη σεβαστούν. Και γι' αυτό καταψήφισα αυτό το ψήφισμα, όχι λόγω του περιεχομένου του, αλλά λόγω του ότι το ψήφισμα αυτό υπάρχει εν πλήρη παραβάση ε, της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Ευχαριστώ κύριος Ζαράντιλ. Ζαχράντιλ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Τι μας ενδιαφέρει. Το Κοινοβούλιο έκανε λάθος σήμερα υπερψηφίζοντας το παρόν ψήφισμα για την κατάσταση στην Πολωνία. Τι έκανε λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, κλάδεψε και πριώνησε το κλαδί στο οποίο κάθεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η πολλαπλή φορά ε, που ε, αναμίχθηκε στα εσωτερικά μιας χώρας ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η τρίτη φορά πρώτα η Αυστρία, μετά η Ουγγαρία, ακολούθησε η Πολωνία και πάντα οι λόγοι ήταν πολιτικοί και τα μέτρα πάντα στρέφονται κατά της κυβέρνησης μιας χώρας που δεν συμμερίζεται με την πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δηλαδή αυτά που φρονούν το ΕΛΚ και οι σοσιαλιστές και δημοκράτες. Τώρα δηλαδή βγάζει μια κίτρινη κάρτα στην πολωνική κυβέρνηση και την προειδοποιεί. Όλα αυτά είναι απαράδεκτη θέματα. Ως μέλος του, της ομάδας μου που έχουμε και την πολωνική ομάδα είμαστε κατά. Η κυρία Μορβάη, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι είναι σπάνιο να μιλάει κανείς σε κενά έδρανα για τόσο σημαντικά θέματα. Και παίρνουμε αποφάσεις και όσοι μας βλέπουν αυτή τη στιγμή και μας παρακολουθούν από το διαδίκτυο θα διαπιστώσουν ότι έχουμε καμιά ντουζίνα βουλευτές παρόντες. Οι Πολωνοί συνάδελφοι τα είπαν πολύ ξεκάθαρα. Ζητήσαμε γραπτός και παρανόμως η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναμειγνύεται στην Πολωνία. Εμείς λέμε με ποια δικαίωμα και με ποια νομική βάση. Το έχουμε ξαναδεί αυτό στην Ουγγαρία. Το κάνανε ξανά και δεν μπόρεσαν να μας πούνε ποια είναι η νομική βάση. Ούτε προθεσμίες στηρίθηκαν, Αντί για έξι εβδομάδες ε, ε, χρειάστηκαν τρεις μήνες για την απάντηση κτλ. Παρακαλούμε λοιπόν τους Ευρωπαίους συναδέλφους να κοιτάνε τα δικά τους προβλήματα ε, και να κοιτάνε τις, τους λαούς στο Βέλγιο και στη Γερμανία. Ας πούμε με βάση ποια νομική διάταξη δέχεστε μαζικά τους μετανάστες παρά τη θέληση του πληθυσμού. Τι χώρες είναι αυτές που δεν λειτουργούν η αστυνομία, οι κρατικές αρχές, για να μην μιλήσω για τις μυστικές υπηρεσίες. Δεν είναι η Ουγγαρία, ούτε η Πολωνία, το Βέλγιο είναι μια τέτοια χώρα. Όπου απέτυχε εκτρά το κράτος δικαίου, δεν υπάρχει κράτος και υπάρχει τρομοκρατία. Λοιπόν, καθίστε στα αυγά σας και ασχοληθείτε με τα δικά σας προβλήματα. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, για... μιλήσατε για ένα λεπτό και 47, ενώ είχατε ένα λεπτό στη διάθεσή σας. Διπλωσιάστε το χρόνο, δεν είναι δυνατόν. Ο κύριος Ζόλτεκ, παρακαλώ, για ένα λεπτό. Ε, οι δράσεις της πολωνικής κυβέρνησης είναι σωστή, όμως ορισμένα σημεία όπως ε, το χάρη η νομοθεσία περί εποπτείας ε, είναι κάτι φρικτό που φαίνεται να έρχεται από τον κομμουνισμό. Όμως, ε, από ό,τι φαίνεται, κάποιοι διθήκονται από τις σοσιαλιστικές δραστηριότητες. Το ψήφισμα ασκεί κριτική για το πώς επιλέχθηκε το συνταγματικό δικαστήριο. Εγώ καταψήφισα αυτό το ψήφισμα, κυρίως γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να παρεμβαίνει στα εσωτερικά μιας άλλης χώρας. Ο Ρόμπερ Σούμαν, ο ιδρυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μάλλον θα στριφογυρίζει στον τάφο του, καθώς θα βλέπει ότι η ωραία ιδέα της κοινότητας των εθνών γίνεται ένα δημιούργημα άσκησης εξουσίας επάνω στους υπόλοιπους και πρόθεσης και της ομοφιλοφιλίας. Ευχαριστώ κύριος Γιούρεκ και εσείς ένα λεπτό. Ευχαριστώ. η Πολωνία, μια χώρα όπου παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, ουσιαστικά δείχνει σήμερα την πολυμορφία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα διάφορα εθνή της Ευρώπης. το χάρη, σήμερα έχουμε μία γιορτή στην ε, Πολωνία και εσείς μας στέλνετε ως δώρο αυτό το ψήφισμα. Πρόκειται για μία μέρα κατά της Πολωνίας. Είδαμε πώς φερθήκατε στο παρελθόν κατά της Ουγγαρίας. Δεν έχει νόημα κάτι τέτοιο. Το άρθρο 7 είναι σαφές και λέει ότι πρέπει να εφαρμόσουμε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά αν συνεχίσουμε με αυτό, θα, έτσι, θα είναι η αρχή της κατάρρευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εσείς θα αποφασίσετε αν αυτό θέλετε να τελειώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι. Ο κύριος Μάμικινς, παρακαλώ. Τελευταία παρέμβαση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Προφανώς, κάθε κυβέρνηση, ε, δημοκρατικά εκλεγμένη πάντα, έχει το δικαίωμα να κάνει μεταρρυθμίσεις. Ιδιαίτερα όταν ο λαός της χώρας το επιθυμεί. Αυτό συμβαίνει και στην Πολωνία. Ακριβώς αυτό. Πλην όμως θα πρέπει και κάθε κυβέρνηση να ακολουθεί και να σέβεται τις συμφωνίες που έχει συνάψει η χώρα στο παρελθόν. Το κράτος έχει συνέχεια. Σήμερα υπάρχουν τεράστια προβλήματα με το κράτος δικαίου, με την ανεξαρτησία των μέσων μαζικής επικοινωνίας και όλα αυτά συνιστούν βασικές και θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό εγώ απήχα στην ψηφοφορία και πιστεύω ότι οι Πολωνοί προσπαθούν να πιέσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και το αντίθετο και προσπαθεί ο καθένας να δει ποιος θα υποχωρήσει πρώτος. Αυτή ήταν η τελευταία παρέμβαση. Ολοκληρώνουμε εδώ τις επεξηγήσεις ψήφου. Διακόπτουμε μέχρι τις 3. Σας ευχαριστώ. <laughs> για